Ο κύριος Αμιάτ Μπασίρ απεχώρησε από την ομάδα EFDD και έγινε μέλος της ομάδας ECR από τις 23 Ιανουαρίου. Τρέχοντος. Να περάσουμε